θεωρούμε ότι με τον τωρινό κανονισμό τα πράγματα θα διορθωθούν όχι γιατί γίναμε πιο έξυπνοι μετά από 8 χρόνια απλώς γιατί μεσολαβεί η εμπειρία που μας διδάσκει πολλά έχουμε το ψήφισμα για αυτό το σημείο και θα ψηφιστεί αύριο επόμενο σημείο έκθεση Πέτερλε σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη δράση κατά του καρκίνου Ευρωπαϊκή Σύμπραξη. Για τέσσερα λεπτά ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι. Με την έκθεση αυτή τοποθετούμαστε πολιτικά σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ο καρκίνος ε, εξαπλώνεται και ένα στους τρεις πολίτες κινδυνεύει. Εγώ χαίρομαι για το ότι στην αρχή αυτής της θητείας δεν χρειάζεται να ζητήσουμε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να κάνουν τα βασικά βήματα γιατί έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2008 και ένα φιλόδοξο σχέδιο της ε, Κομισιόν που ονομάζεται «Καταπολέμηση του καρκίνου» και αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης. Είναι σημαντικό το ότι αναλαμβάνουμε ήδη δράση και υποστηρίζουμε έτσι ένα σημαντικό φιλόδοξο στόχο της Κομισιόν, δηλαδή να μειωθεί σε 10 χρόνια 10% να μειωθούν τα κρούσματα καρκίνου. Επίσης χαίρομαι για το ότι αυτό έγινε σύμφωνα με το ψήφισμά μας για τη στρατηγική υγείας μαζί με την ε, περίοδο 2008-2013. Λέμε εδώ πέρα στο ψήμα πως πρέπει να βοηθήσουμε στην υγεία για όλους και να δοθεί η έμφαση στην ε, πρόληψη. Είναι πολύ ανησυχητικό το ότι κατά μέσο όρο οι χώρες επενδύουν μόνο 3% του υπερβολισμού υγείας στην πρόληψη. Δηλαδή φαίνεται σαν στατιστικό λάθος, αλλά φαίνεται πως δεν συμπεριλαμβάνεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό η πρόληψη. Πρέπει να αλλάξουν εδώ πέρα τα πρότυπα λοιπόν, να επενδύσουμε σε στρατηγικές προσεγγίσεις οργανωτικές και τεχνολογικές. Έχει αποδειχθεί πως η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μειώνει την θνησιμότητα. Επίσης, άλλο σημαντικό κομμάτι, η ανισότητα. Υπάρχουν πολλά είδη ανισότητας εδώ πέρα. Το σημαντικότερο είναι το αυτό το οποίο λέμε το σιδηρούν παραπέτασμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στις ε, πιθανότητες επιβίωσης όσων ασθενών από καρκίνο αλλά και εντός των κρατών μελών. Υπάρχουν διαφορές στο ποσοστό επιτυχίας παρέμβασης ε, και αντιμετώπισης ε, του καρκίνου, επίσης το τι γίνεται με την επανένταξη των ασθενών οι πολίτες ε, της Ένωσης δεν ε, ξέρουν καν ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Κάποια κράτη-μέλη έχουν εθνικά προγράμματα, αλλά δεν έχουν καν. Υπάρχουν επίσης διαφορές στην ε, συλλογή στατιστικών δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο την δυνατότητα μέτρων στήριξη σύμφωνα με τις συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση σε αυτό το επίπεδο. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών δεν θα γίνει αν δεν την υποστηρίξουν τα θεσμικά όργανα. Τρίτο κομμάτι, συνεργασία. Ο φιλόδοξος στόχος της Κομισιόν θα επιτευχθεί μόνο εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τρόπο κάθτο και οριζόντιο βασική προϋπόθεση εδώ πέρα είναι ο καρκίνος να συνεχίσει να μας απασχολεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι στενές σχέσεις μεταξύ ασθενών και ιατρών δεν αρκούν. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε σε μια πολιτική συνεργασία, σε πολιτική θέληση που θα δώσει μια άλλη δυναμική σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα θα ήθελα να τονίσω την σημασία επανένταξης των καρκινοπαθών. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με όσους βγαίνουν νικητές από τη μάχη με τον καρκίνο. Δεν πρέπει να υπάρχει στίγμα ή να τους ξεγράφουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να επανεντάσσονται στην κοινωνική ζωή και να έχουν τη δυνατότητα να επανταχθούν στην προηγούμενη του σταδιοδρομία. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ηγητές ε, και όλους όσους με βοήθησαν. Το λόγο, το λόγο έχει ο Επίτροπος Νταλή. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, χαίρομαι διότι είσαστε ενθουσιώδεις και υποστηρικτικοί ως προς την εργασία μας για τον έλεγχο του καρκίνου. Χαίρομαι για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ιδιαίτερα από τον εισηγητή, τον κύριο Πέτερλε. Χρειάζεται δυνατή δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να υπογραμμίσουμε την εταιρική σχέση και υποστήριξή μας όλα εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή, συμμετοχή των διαφόρων εταίρων. Μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη, η υπεύθυνοι τομέα υγείας, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φαρμακοβιομηχανίες έχουν συμμετάσχει σε συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του 2013. Θα πρέπει να δούμε όμως κατά πόσο αυτά τα νέα μέσα συνεργασίας θα οδηγήσουν σε βιώσιμη συνεργασία αντιμετώπισης του καρκίνου. Ελπίζω αυτή την πορεία να ακολουθήσουμε. Οι ευρύτεροι στόχοι για, μακρόπνοους, για αποτελέσματα σημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση πόρων και μέσων. Και βεβαίως ε, αυτό σημαίνει επαρκή χρηματοδότηση. Θα πρέπει να ενταχθούν, να εγγραφούν νέα κονδύλια σε μελλοντικούς προϋπολογισμούς. Μιλάμε για μία εκτενή προσέγγιση πρόληψης και αντιμετώπισης καρκίνου. Πολλά μέτρα ελήφθησαν υπόψη στα πλαίσια της εταιρικότητας. Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής έχουμε πέντε πυλώνες στην πρόληψη, και την πρόθεση του Ευρωπαϊκού ε, Κώδικα κατά του καρκίνου, παρακολούθηση και προσυμπτωματικός έλεγχος, ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών στην αντιμετώπιση του καρκίνου, συνεργασία και συντονισμός έρευνας κατά του καρκίνου και συγκρίσιμες, ε, συγκριτικές πληροφορίες και δεδομένα για τον καρκίνο έτσι ώστε να βελτιώσουμε τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια κατά του καρκίνου. Στο τέλος του εταιρικού σχεδίου θα πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα από όλα τα κράτη-μέλη με βάση και την έμπρακτη μέχρι τούδε εργασία. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να προβάλλει κάθε υποστήριξη και θα συνεχίσουμε σε στενή συνεργασία στην, με, την, με το Διεθνή Οργανισμό Καταπολέμησης του Καρκίνου. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη ενσωμάτωση συνιστοσών υγείας σε όλα τα εθνικά μας προγράμματα. Και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την πρόληψη για να καταπολεμήσουμε έμπρακτα τον καρκίνο. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουμε και αναμένω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Περνάμε στις ομάδες εξ ονόμαστος των σοσιαλιστών. Έχει το λόγο ο κύριος Παρνιό. Κύριε Πρόεδρε κύριε Νταλή. Η έκθεση του κυρίου Πέτερλε λαμβάνει υπόψη της την έκθεση της Κομισιόν αλλά και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ου του 2008 για την καταπολέμηση του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να υποστηρίξω τους στόχους για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη στην καταπολέμηση του καρκίνου και τονίζω ότι χρειάζεται πρόληψη, επεξεργασία ενός νέου μοντέλου ε, για την πρόληψη και μείωση των ασυνοτήτων μεταξύ κρατών μελών. Σημερίζομαι αυτά τα οποία λέει η Κομισιόν και χαιρετώ, χαιρετίζω την εργασία του κυρίου Πέτερλε. Και κυρίως για να βρεθεί ο συμβιβασμός τον οποίο πετύχαμε. Θα ήθελα να τονίσω εγώ ως εισηγητής της σοσιαλιστικής ομάδας τα εξή αύξηση των θανάτων από καρκίνο λόγω έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας, βελτίωση της φαρμακολογίας ε, για τους ε, αρρώστους ε, από καρκίνο, συμπλήρωμα του ρίτσα, απαγόρευση εισαγωγή εμπορευμάτων με καρκινογόνες ουσίες, απαγόρευση δε της χρήσης αυτών των ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης ε, σταμάτημα των εμποδίων για την ε, ε, κοινωνική ζωή των ανθρώπων με αρρώστιες. Η κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πέτερλε για την εξαιρετική του εργασία, έτσι ώστε η καταπολέμηση του καρκίνου να αποτελέσει ε, υψηλή μας προτεραιότητα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα αριθμητικά στοιχεία. Ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα δραστικά. Το, ο φόρτος του καρκίνου αποτελεί απειλή για τα εθνικά συστήματα υγείας και θα πρέπει να ανταποκριθούμε επαρκώς όταν μιλάμε για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, μιλάμε για εταιρικότητα. Αλλά θα καταπολεμήσουμε τον καρκίνο αν είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ιδιαίτερα οι ασθενείς συμμετέχουν ενεργά με τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Και βεβαίως με την παρακολούθηση αυτής της εταιρικής σχέσης ελπίζω η Επιτροπή να διαδραματίσει το σωστό ρόλο έτσι ώστε η εταιρικότητα αυτή να αποδώσει. Θα ήθελα η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το υπάρχον ECDC. Αυτό θα βελτιώσει την πραγματογνωμοσύνη μας έτσι ώστε να έχουμε έγκαιρη ε, προσπελασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταπολέμησουμε τον καρκίνο μέσα στα πλαίσια ενός απότερου στόχου. Την μείωση των ε, ανισοτήτων ε, υγείας στην Ευρώπη και θα ήθελα αύριο κύριε Επίτροπε να συμμετάσχετε στην ημερίδα καταπολέμησης των νόσων. Από την ΚΟΕ. Για ένα λεπτό. Η κυρία Λεωτάρ. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και κύριε Σίγητα. Είναι μια τρομακτική ασθένεια ο καρκίνος Και ισχυρότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Αλλά ευτυχώ εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ζούμε περισσότερο χρόνο, οπότε δυστυχώ είναι μεγαλύτερο ο κίνδυνος καρκίνο. Όσο πιο ηλικιωμένο ο πληθυσμό, τόσο πιο περισσότερα κρούσματα. Γι' αυτό πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να βρουν μια στοχευμένη πολιτική υγείας και με προληπτικό έλεγχο και με αντικαρκυνικά φάρμακα τα οποία θα μπορεί να πληρώσει ο κόσμος. Επίσης ε, θα, πρέπει να εξασφαλίσουμε τις καρκινογόνες ε, ουσίες από το περιβάλλον, από τις ε, οικίες μας. Σκεφτείτε μόνο τον αμίαντο. Ακόμα και αν χρειαστεί να βλάψουμε κάποια ε, βιομηχανικά συμφέροντα, καθώς σημαντικότερο είναι ο υγιής πολίτης. Σας ευχαριστώ για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για ένα λεπτό η κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε πως είναι μαζική η ασθένεια πλέον, ξέρουμε πως μπορεί να υπάρχει βεβαίως και γενετική ε, προδιάθεση και να ε, αποκτήσει κανείς καρκίνο από... Πρόκειται για μια φρικτή αρρώστια η οποία πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους και έχουμε πάρα πολλούς θανάτους εγώ χαίρομαι για αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα για την καταπολέμηση του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ τώρα τι, ποια είναι η θέση της Κομισιόν για την έρευνα. Μπορείτε να προβλέψετε κονδύλια για να διασφαλίσετε την έρευνα. Ποια είναι η προτεραιότητα που της δίνετε. Επίσης, πώς θα υλοποιήσετε αυτά τα φιλόδοξα σχέδια. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητες πρόληψης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Θανασέσκου για 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτερλε για τη δουλειά του. Τα ιατρικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο καρκίνος είναι και ο πρώτος λόγος θνησιμότητας στην Ευρώπη. Αυτή η πρόταση για σύμπραξη στην καταπολέμηση του καρκίνου είναι μια εξαιρετική ιδέα και για τους αρρώστους αλλά και για τις οικογένειές τους. Η συνεργασία πρέπει να είναι συνεχής και μόνιμη για να μπορέσουμε να βρούμε και τις λύσεις. Πρέπει η ευρωπαϊκή συνεργασία για την καταπολέμηση του καρκίνου να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα τα κονδύλια, το know-how και τις δυνατότητες των κρατών μελών, τις υποδομές. Και όλη η ερευνητική βιβλιογραφία που υπάρχει στα κράτη-μέλη πρέπει να διατίθεται και στα άλλα κράτη-μέλη. Η κυρία Εστρέλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η καταπολέμηση του καρκίνου θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Το 30% των καρκίνων μπορούν να αποφευχθούν με βάση τον ε, προληπτικό έλεγχο. Ε, ορισμένοι τύποι καρκίνου πλήττουν διαφορετικά άνδρες ή γυναίκες. Έχουμε 275.000 γυναίκες ετησίως με καρκίνο του μαστού και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες. η γυναικες εχουμε 275000 γυναικες ετησιως με καρκινο του μαστου και αυτο το βλεπουμε ιδιαιτερα στις νεες γυναικες ο καρκίνος του καρκίνου πλήττει 50.000 γυναίκες ετησίως και 25.000 γυναίκες πεθαίνουν. Μπορούμε όμως να αποφύγουμε τον καρκίνο του καρκίνου με βάση το, ένα συγκεκριμένο εμβόλιο. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι γυναίκες να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο με βάση συγκεκριμένες εκστρατείες υγείας και με βάση την έγκαιρη διάγνωση έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουμε ποια είναι τα υπάρχοντα προγράμματα πρόληψης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στρέλα. Η κυρία Αντωνέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή στην, στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν ανακοινώνει ότι ο αριθμός των τεστ πρόληψης στην Ένωση είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού. Πρέπει όμως να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό, διότι και η ακρίβεια των ε, τεστ έχει αυξηθεί και είδαμε και στο ιατρικό σαλόνι της Γενέβης ε, ένα μηχάνημα μίας Ρουμάνας ερευνήτριας που επιτρέπει ανείχνευση του καρκίνου μέσα σε έξι λεπτά. Η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών πρέπει να ενδιαφερθούν για την, την εφεύρεση και να την συμπεριλάβουν στις κατευθυντήριες γραμμές. Ο κύριος Λούαν με τη μέθοδο του Κατζδεάη. είναι απαραίτητο αυτό το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου που είναι η δεύτερη αιτία θνησιμότητας στην Ευρώπη. Υπάρχει όμως μια μεγάλη ανισότητα μεταξύ κρατών μελών για την ποιότητα της θεραπείας και την πρόσβαση. Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης υπάρχει <laughs> υπάρχουν δύο φορές, μάλλον στη Νότια Ευρώπη το ποσοστό θνησιμότητας είναι το διπλό από ό,τι στην ε, Βόρεια Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε εμεί αυτές τις ανισότητες. Πρέπει η Κομισιόν να χρηματοδοτήσει την έρευνα. Η ρουμάν επιστημόνισσα που ανακάλυψε αυτό το τεστ ανείχνευσης πρέπει να χρηματοδοτηθεί όπως και η αντίστοιχη έρευνα που γίνεται. Με αυτό το μηχάνημα με λιγότερα από 6 λεπτά ανοιχνεύει κανείς το καρκίνο. κυρία Σίλροβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ακούστηκε πως η αποτελεσματική καταπολέμηση του καρκίνου πρέπει να περιέχει πολλά πράγματα από την αναγνώριση μέχρι την περίθαλψη. Πρέπει όμως να πούμε το εξής. Υπάρχουν και οι οικογένειες των ασθενών που χάνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Πρέπει να τις ε, ενθαρρύνουμε, αλλά βεβαίως απέναντι σε αυτή την αρρώστια είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν πρέπει λοιπόν να μένουν μόνες τους οι οικογένειες όταν μιλάμε για καταπολέμηση του καρκίνου. Πρέπει να σκεφτούμε και τους συγγενείς αυτούς. Η βοήθεια λοιπόν σε αυτές τις οικογένειες δεν πρέπει να γίνεται μόνο κατοικών αλλά να υπάρχει και πρόσβαση σε ειδικά νοσοκομεία που θα βοηθήσουν αυτούς τους ασθενείς μέχρι το τελευταίο στάδιο. Ευχαριστώ. κύριος Γκάλαχερ έχει τον λόγο, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπολογίζεται πως 3,2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ε, διαγνώσκεται ότι έχουν καρκίνο κάθε χρόνο και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις τάσεις αυτές οι διαγνώσεις θα διπλασιαστούν τα επόμενα 20 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να δούμε την πληγή, τη μάστιγα αυτού του καρκίνου που προκαλείται από πολλούς ε, παράγοντες π.χ. το κάπνισμα, το να είναι κανείς η ε, υπέρβαρος, ε, η μικρή κατανάλωση λαχανικών, Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τις στρατηγικές υγείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στους πόρους και σημαντική είναι η εγκαιρή διάγνωση και βλέπουμε πως η διάγνωση είναι τόσο σημαντική καθώς ζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα ζούσαν διαφορετικά. Μέσω της έρευνας αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα ηγετικό ρόλο πάνω από 750 εκατομμύρια έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή για την έρευνα του καρκίνου υπό το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ελπίζω πως θα έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια και θέλω τέλος να αναφέρω όλους όσους ειδικά από τη χώρα μου φροντίζουν τους καρκινοπαθείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βέρμπερ τώρα έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η υγεία βεβαίω είναι ένα αγαθό που πρέπει να διαφυλάξουμε. Ο καρκίνο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται το 2004 σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΠΟΕ 13% όλων των θανάτων οφείλονταν σε αυτό. 3,2 εκατομμύρια κρούσματα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κάθε χρόνο με κύριες περιπτώσεις των καρκίνο των πνευμόνων και του στήθους. Θεωρούμε λοιπόν ότι η καλύτερη στρατηγική με την υψηλότερη επιτυχία είναι η διάγνωση και η πρόληψη. Σας ευχαριστώ κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι πρέπει να δούμε τι γίνεται με την έρευνα στον καρκίνο και στη δική μου τη χώρα πεθαίνουν νέοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι κάθε μέρα και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως ένας στους τρεις ανθρώπους θα μπορούσε να επηρεαστεί από τον καρκίνο. Ταυτόχρονα σημειώνεται μεγάλη πρόοδος ε, γίνεται δουλειά από γιατρούς και ασθενείς για την αντιμετώπιση αυτής της ε, ασθενής και τις νοσοκόμες και τους νοσηλευτές και πρέπει λοιπόν να αφιερώσουν περισσότερα χρήματα στην έρευνα και εδώ είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέσει κονδύλια για την έρευνα πρώτα απ' όλα και να υποστηρίξει τη συνεργασία με τα Ινστιτούτα εκείνα τα ερευνητικά. Εάν το κάνουμε αυτό θα έχουμε περισσότερη πρόοδο στο μέλλον και λιγότεροι άνθρωποι θα αρρωστιένουν. Σας ευχαριστώ κυρία Μορβάη kérek, egy kicsit a szokásosnál személyesebb. Ευχαριστώ. Λυπάμαι γιατί μιλώ πιο προσωπικά από το σύνηθες, αλλά επειδή μιλάμε για την καταπολέμηση του καρκίνου, όλοι ανέφεραν τον αριθμό των θυμάτων, τον υψηλό αριθμό θυμάτων. Τέσσερα χρόνια πριν και εγώ αντιμετώπισα αυτή την ε, ασθένεια έπρεπε να δώσω μεγάλη μάχη και ακολούθησα χημειοθεραπείες πολλές εβδομάδες. Σήμερα βρίσκομαι εδώ, είμαι ευρωβουλευτής, έχω τρία παιδιά και μπορώ να ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω έκκληση προς όλους τους ε, πολίτες να προβαίνουν σε προσυμπτωματικό έλεγχο και θα ήθελα να παρεκτείνω τη σκέψη μου σε αυτούς που νοσούν, να μην χάνουν ποτέ την ελπίδα τους. Ευχαριστούμε, κυρία Μορβάη. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος ε, με τον ενθουσιασμό που κατέδειξε το Κοινοβούλιο σήμερα ως προς το μεγάλο θέμα της ενιαίας καταπολέμησης αυτής της νόσου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτερλε, τον εισήγητη, για την πραγματική του συνεισφορά και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μόρβάη ιδιαίτερα που μας μίλησε για την θετική πλευρά της ελπίδας. Δεν χάνονται όλα ενώπιον αυτής της ασθένειας. Πολλά σημεία εθίγησαν, πολλές απόψεις εκφράστηκαν Προσδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτά που είπατε και αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση της Κομισιόν και θα ήθελα να σας εγγυηθώ ότι οι σημερινές παρεμβάσεις θα μελετηθούν διεξοδικά προγραμματίζοντας τις μελλοντικές μας δραστηριότητες. Ως προς τους ε, περιβαλλοντικούς παράγοντες, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το περιβάλλον είναι καθοριστική σημασίας για την καταπολέμηση του καρκίνου. Όμως, οι υψηλές προδιαγραφές που διαθέτουμε στην Ευρώπη υποβοηθούν την ε, φθήνουσα σημασία αυτής της νόσου. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε υψηλές ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Τώρα, ως προς την έρευνα και η έρευνα θα πρέπει να μας απασχολήσει. Οι φαρμακοβιομηχανίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και κατέχουν σημαντική θέση στη γενική μου διεύθυνση και έχουμε μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας με την ε, φαρμακευτική βιομηχανία για να συντονίσουμε καλύτερα τις ερευνητικές μας δραστηριότητες και για να εγγυηθούμε την καλή λειτουργία της έρευνας αυτής. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της, δραστηριότητας μου, της δραστηριότητάς μου είναι ε, να εγγυθώ την προσβασιμότητα, την προσπελασιμότητα για τα φαρμακευτικά σκευάσματα στην αγορά, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρώπη σήμερα είναι η ανισότητα, οι μεγάλες ανισότητες πρόσβασης στα συστήματα υγείας. Αυτό θα πρέπει να το εγγυηθούμε με βάση την καλύτερη προσπελασιμότητα στα φάρμακα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα εν κατακλείδη να πω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας έτσι ώστε να πείσουμε τους πολίτες για τη σημασία της πρόληψης του προσυμπτωματικού ελέγχου. Μιλήσαμε για τον καρκίνο του μαστού. Έχουμε την δυνατότητα screening και οι γυναίκες θα πρέπει να υφίστανται ε, τακτικούς ε, προσυμπτωματικούς ελέγχους. Ο κύριος Πέτερλε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η απόψινή συζήτηση ήταν πραγματικά ευχάριστη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι που μιλάμε την ίδια γλώσσα και έχουμε τους ίδιους στόχους. Νομίζω πως συμφωνούμε όλοι ε, για το ευρύτερο πλαίσιο και για τους λόγους ε, εδώ πέρα, αλλά χρειαζόμαστε και αυτή τη συνεργασία. Πριν δεν είχα αρκετό χρόνο για να πω κάποια λόγια για την υγιεινή ζωή. Είμαι πεπισμένος πως μπορούμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα εδώ πέρα και εμείς οι πολιτικοί δίνοντας το καλό παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τον υγιεινό τρόπο ζωή Εγώ ο ίδιος. Ε, είχα και εγώ μια ανάλογη διάγνωση όπως η κυρία Μορβάη την οποία θέλω να συγχαρώ καθώς έτσι αποδεικνύουμε πως ο καρκίνος δεν σημαίνει απαραίτητα θανατική καταδίκη. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, να τον ευχαριστήσω που ανακοίνωσε ε, επιτάχυνση της δραστηριότητας σε αυτόν τον τομέα. Ο καρκίνος είναι πολύ δυναμική, αλλά και το ίδιο πρέπει να ε, είμαστε και εμείς ε, και ναι, όπως ελπίζω και στο μέλλον να συνεχιστεί η υποδεγματική συνεργασία που έχουμε. Να πω επίσης σύντομα πως θα ξανασυσταθεί μια ομάδα που λεγόταν MAG, δηλαδή βουλευτές κατά του καρκίνου. Νομίζω τώρα πως με τη νέα ομάδα θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη. Σας ευχαριστώ όλους και καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε κύριε Πέτερλε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι